έχω μια υποβολή αίτηση για ένα διορισμό σε μια επιτροπή και θα δημοσιευθεί στα πρακτικά αυτή τη συνεδρίαση. Και εφόσον ε, δεν υπάρξουν